Well, hello everyone. You have received Λοιπόν, λάβατε την ημερήσια διάταξη και αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Έχω μερικές ανακοινώσεις να σας κάνω. Λάβαμε από το Συμβούλιο διορθωτικά το ένα για τον κανονισμό για τις ε, ιατροτεχνικές συσκευές και το δεύτερο για τον κανονισμό για τη διάγνωση in vitro και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγξει αυτά τα κείμενα και να τα εγκρίνει. Στις 20 Μαρτίου, χτες, ε, λάβατε αυτά τα κείμενα και η προθεσμία λήγει σήμερα. Δεν έχω λάβει κανένα αίτημα για αλλαγή, οπότε μπορώ να σας ανακοινώσω τώρα ότι εγκρίνονται τα δύο αυτά διορθωτικά από την Επιτροπή μας και θα αποσταλούν στις υπηρεσίες της Ολομέλειας για να ανακοινωθούν αντιστοίχως και να εγκριθούν και από την Ολομέλεια. Στο φάκελο σας επίσης έχετε τις εκθέσεις της αποστολής στην COP24 στο Κάτω Βίτσε, στο Νέι Μέχεν της Ολλανδίας. Είναι ευρωπαϊκή πράσινη πρωτεύουσα και αποστολή στην Κίνα για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Αυτές ήταν οι ανακοινώσει που είχα να σας κάνω. Θα ήθελα να σας θυμίσω δε ότι την άλλη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα κάνουμε δεξίω την Τετάρτη. Έχω στείλει σε όλους ε, προσκλήσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε αν θα έρθει επίτροπος και από το Συμβούλιο, έτσι για να ε, κλείσουμε τη θητεία στις 6 και 4 μετά τις ψηφοφορίες της Τετάρτης. Ελάτε, αλλά παρακαλώ να το δηλώσετε στη γραμματεία. Ε, απαντήστε. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες, όπως βλέπετε, και ως ήθιστε... Έχετε ηλεκτρονικά το φάκελο με τα έγγραφα και η ε, συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδικτύο. Επίσης, έχετε και τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 26 και 27 Φεβρουαρίου. Ε, αν δεν διαφωνήσει κανείς και δεν προπαλεντρήσει μέχρι το τέλος της συνεδρίας, θα θεωρώ ότι εγκρίνονται. Πρώτο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε είναι αντίδραση, αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 για την χρήση ορισμένων μάλλον για ορισμένε χρήσει του τριοξιδίου του χρωμίου. Ο κύριος Έκχαουτ είναι ο εισηγητής, αλλά απουσιάζει και θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Χόισλινγκ, ο οποίος ε, και έχει μέσα στο λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και πάλι πρόκειται για την έγκριση μιας ουσίας που είναι υψηλού κινδύνου, το τριοξίδιο του χρωμίου, ούτε να το πω δεν μπορώ. Είναι καρκινογόνο για τον άνθρωπο και χωρίς οριακές τιμές. Ε, οπότε προβληματικό. Δύο είναι οι προϋποθέσεις. Οι κοινωνικο-οικονομικά ε, λέει πλεονεκτήματα που είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους και δεν υπάρχουν και ασφαλείς εναλλακτικέ προτάσεις. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως τι κάνει αυτή η ουσία, τι συνέπειες έχει. Είναι πάρα πολύ ευρεία η πρόταση έγκρισης. Το τριοξίδιο του χλωρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, σε εξαρτήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, σε κραγιών, ε, σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε στην αεροπορία, ε, σε βρύσες είναι τελείως ε, ασαφή και αόριστα ε, και ε, ποιες θα είναι οι εφαρμογές δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι δεν ξέρουμε. Και ποια είναι η κοινωνικο-οικονομική ανάλυση δεν είναι εφικτή. Δεύτερον, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να εξακριβώσουμε αν υπάρχουν αλλακτικέ λύσεις. Δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις. Το Σεπτέμβριο του 2018 έκανε μια έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι μερική η ενημέρωση. Υπάρχουν μεγάλες ε, ελλείψεις και ασάφειες. Δύο, τι να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, απαγόρευση της έγκρισης, ε, γιατί δεν ε, συνάδει με την ε, νομοθεσία REACH. Και το δεύτερο, να εγκριθεί μετά από έλεγχο ε, της ε, κείμενης νομοθεσίας κατά πόσο μπορεί να είναι ε, δυνατή η συνύπαρξη. Υπάρχει μια απόφαση της 7ης Μαρτίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια να διαπιστώσει αν πληρούνται οι όρικοι προϋποθέσεις. σαν να ζητάς να βγάλεις δίπλωμα οδήγησης και να πεις «Ε, θα σας προσκομίσω στη συνέχεια την οφθαλμιατρική εξέταση. Δώστε μου το δίπλωμα οδήγησης, θα σας φέρω μετά τα στοιχεία και τα παραστατικά που απαιτούνται. Ε, κάτι τέτοιο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη ουσία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κατονομάσει τις εναλλακτικέ ε, λύσεις που δεν υπάρχουν, αλλιώς δεν πληρούν τα κριτήρια για την, ένταξη, για την έγκριση και πάλι αναφέρομαι στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι ακολουθεί την ίδια τακτική να το εγκρίνουμε πρώτα και μετά να φέρουν τα στοιχεία. Υπάρχουν και κάποιες ανασφάλειες και αβεβαιότητες σε σχέση με τις εναλλακτικέ ουσίες. γιατί, τι θέλω να πω με όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την προηγούμενη σε σχέση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Βάσει της απόφασης του δικαστηρίου είναι παράνομη η έγκριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αλλάξει την έγκριση, θα την αρνηθεί ή θα τη φέρει σε ψήφιση. Πρέπει να μας απαντήσει. Κανονικά η μόνη σωστή λύση είναι η απόρριψη. Ξέρουμε ότι το ξασθενές χρώμιο χρησιμοποιείται παντού, πάλι μέχρι, από τα κραγιόν μέχρι τους δορυφόρους. Και μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες μία άρνηση έγκρισης κυλοφορίας του προϊόντος αυτού στην αγορά. Πρέπει να ξέρουμε τι αιτήσει έχουν κάνει, ποιε εταιρείε και ποιες είναι οι συγκεκριμένες εφαρμογές ε, που γνωρίζουμε. Ε, προτείνουμε ένα συμβιβασμό απόρριψη της γενικής έγκρισης για γενική κυκλοφορία και ανεξέλεκτη και έγκριση περιορισμένων ε, εφαρμογών που ανταποκρίνονται στην νομοθεσία REACH. Κατ' εξαίρεση να εγκρίνουμε κάποιες εφαρμογές σε περιορισμένο χρονικό ε, διάστημα για να έρθουν τα επιπλέον δικαιολογητικά και στοιχεία. Επειδή λοιπόν μας έχει απασχολήσει το θέμα του εξασθενούς χρωμίου εκτός από το τριοξίδιο, θέλουμε να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στη βιομηχανία για να διορθώσει τα κακό κείμενα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να σεβαστούμε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλιώς ε, παράνομα θα δώσουμε μια έγκριση για κάτι το οποίο μπορεί να προσβληθεί ενώ ξέρουμε ποιε είναι οι διαδικασίε και θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο αναπεθυμίτες ενέργειες. Δεν υπάρχουν ωριακέ τιμέ. Είπαμε ότι είναι ξεκάθαρα καρκινογόνα η ε, ουσία, το ξέρουμε. Ε, τι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να μείνει έτσι ε, όπως έχει. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τι ευθύνε τη και εμεί να το διορθώσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κωστέτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό θα διαφωνήσω και θα υποστηρίξω την πρόσθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα εξηγήσω και γιατί. Κανεί βεβαίω δεν αμφισβητεί ότι το χρώμιο 6 έχει ε, ε, τέτοιε ιδιότητε καρκινογενεί, ε, ε, αλλά χρειάζεται πολύ αυστηρές προφυλάξει σε ό,τι αφορά τη χρήση του και σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων αλλά και σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή βασίζεται στην γνωμάτευση της Επιτροπής ΕΚΑΜ και θεωρεί ότι οι κίνδυνοι από αυτή την ουσία μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο και μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτή την ουσία όσο δεν έχει βρεθεί μία εναλλακτική η οποία είναι αξιόπιστη. Το χρώμιο 6 είναι απαραίτητο για μια σειρά από βιομηχανικές εφαρμογές και γνωρίζω πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. Διότι αν κάποιες μπορεί να υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια υποκατάστατα και σχετικές διαδικασίες, αλλά έχουν τα όρια τους και δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Η χρήση του τριοξιδίου χρωμίου πλαισιώνεται άλλωστε ήδη σε κάποια, σε κάποια κράτη-μέλη. Στη Γαλλία υπάρχουν προϋποθέσεις χρήσης του προϊόντος αυτού εξαιρετικά αυστηρές. Η γαλλική νομοθεσία προβλέπει οριακές τιμές ε, επαγγελματικής έκθεσης και αυτές οι οριακές τιμές ε, είναι εξαιρετικά χαμηλές. Γιατί λοιπόν να μην ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα. Υπάρχει και το benchmark. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το προϊόν πλαισιώνοντάς το με αυστηρές προϋποθέσεις και χαμηλές οριακές τιμές, ας εκμεταλλευτούμε αυτή την εμπειρία που υπάρχει. Το υπενθύμισε ο προηγούμενος ομιλητής, χωρίς παράταση της άδειας δεν θα μπορούμε στον τομέα της αερονοσπηγικής να επεξεργαστούμε την επιφάνεια κάποιων ε, εξαρτημάτων. Δεν θα μπορεί πια να γίνει αυτό στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει η επεξεργασία εκτός Ευρώπης και μετά θα τα επανεισάγουμε. Οπότε σκεφτείτε λίγο και τις επιπτώσεις για τον του άνθρακα. Και θα έχουν επεξεργασμένα ε, προϊόντα τα οποία θα μπορούν να κυκλοφορούν στην Ευρώπη χωρί περιορισμού. Και αυτό βεβαίω θα πλήξει όχι μόνο την αγωνιστικότητα τη βιομηχανία μα, αλλά θα μετατοπίσει το πρόβλημα σε κάποιε περιοχέ του κόσμου όπου η περιβαλλοντική και η υγειονομική νομοθεσία προστατεύει πολύ λιγότερο. Εάν δούμε λοιπόν τη σχέση ε, κινδύνου-οφέλους, ε, της χρήσης του, του τριοξιδίου του χρωμίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ε, δεν νομίζω να πρέπει να αμφισβητήσει κανείς την ομάδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ την κυρία Γκροστέτ και τώρα ο κύριος Μπαλέτ. Μπέλετ. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Τα πιο σημαντικά στοιχεία ήδη τα ανέφερε η Φρανσουάζ. Απλώς να προσθέσω και εγώ κάποια στοιχεία. Καταρχάς, η Φρανσουάζ αναφέρθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το αίτημα για την έγκριση της λάξης ε, έχει υποστηριχθεί από 150 χρήστες που ε, ε, χρειάζονται το τριοξίδιο του χρωμίου. Αυτοί πήραν την πρωτοβουλία να υποβάλουν αυτή την αίτηση και δεν είναι απλό κάτι τέτοιο, γιατί υπήρχε πολύ διοικητικό άχθος, φόρτος, εργασίε για να το κάνουν αυτό. Οι μεγάλες εταιρείε ήδη έχουν πάρει έγκριση για να το χρησιμοποιούν το τριοξίδιο. Και μάλιστα σε πολλέ περιπτώσει για δωδεκαετία. Άρα, η έγκριση, το αίτημα για έγκριση που εξετάζουμε εδώ αφορά κυρίω. Είναι περιορισμένο μάλλον στο χρόνο 4-6 χρόνια. Με σαφή όρια και σαφή ρήτε αναθεώρηση, όπω ανέφερε και η Φρανσουάζ. Ε, να σχολιάσω την έκθεση τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Διότι αν διαβάσετε το κείμενο τη αντίρρησης φαίνεται πραγματικά να είναι κάτι το τρομερά απειλητικό από την πλευρά της υγείας. Όμως, αν διαβάσετε το κείμενο τη Συμβουλευτική Επιτροπής, λέει ότι οι αναφορές στον αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, όπως ανέφερε δεν ισχύουν. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, οι επιστήμονε δηλαδή οι ίδιοι, λένε ότι ο συνολικό αριθμό ε, κρουσμάτων που εντοπίστηκαν από όσου υπέβαλαν την αίτηση έχουν υπερεκτιμηθεί. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Και τελευταία πρόταση λέει έτσι η ε, χρήση αυτών των εκτιμήσεων που χρησιμοποιούν εδώ και όσοι προβάλλουν αυτή την αντίρρηση, εκτός μιας συγκεκριμένης ε, κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης, δεν ενδείκνυται. Άρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτό του ευρύτερου συγκεκριμένου πλαισίου. Αυτό κάνουν όσοι υπέβαλαν την αντίρρηση. Μιλάμε για εναλλακτικά ε, αποδεκτικά στοιχεία που χρησιμοποίησαν συντάκτε τη αντίρρηση. Το δεύτερο στοιχείο, και το ανέφερε η Φρανσουάζ, τι ενδεχόμενε εναλλακτικέ, όταν υπάρχουν, για προϊόντα που θα έπρεπε να είναι αυλαβή, να τα χρησιμοποιούμε. Και εδώ η Συμβουλευτική Επιτροπή λέει ότι συμφωνεί. Συμφωνεί μετά από μια αξιολόγηση και συμφωνεί ότι η χρήση των εναλλακτικών δεν προλαβαίνει να γίνει εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. Είναι πιο περίπλοκο το κείμενο τους. Και μετά το τελευταίο στοιχείο, αναπομπή στο... στην απόφαση του δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου θα μπορούσε να υπάρξει μια παράλληλη εξέταση, αλλά δεν είναι σαφές ότι θα γίνει αυτό και πραγματικά α δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξετάσει το θέμα σε όλε τι λεπτομέρειε για να δει το πώς ε, επηρεάζει η απόφαση του δικαστηρίου. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία Οποιαδήποτε έγκριση που είναι αντικείμενο αντίρρηση ένσταση ή μορφή από οποιοδήποτε, το ανέφερε και η Φραντσουάζ, μπορεί να μετατοπιστεί απλώ η παραγωγή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση με λιγότερο έλεγχο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην είμαστε αφελεί και πάρουμε αυτόν τον κίνδυνο, αν διατρέξουμε αυτόν τον κίνδυνο. Εδώ Ξέρουμε πόσο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και να ελέγχουμε το προϊόν, αλλά η έγκριση δεν αφορά την έγκριση που ήδη έχει δοθεί για 12 χρόνια στις μεγάλες εταιρείε. Μιλάμε για ε, συγκεκριμένη στο χρόνο ε, έγκριση με συγκεκριμένα ανώτατα όρια και συγκεκριμένη ρήτρα θεώρησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό δεν συμφωνούμε με την αντίρρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο για το θέμα. Εάν όχι, ο κύριος Φίε από την Επιτροπή. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Σημειώνουμε τις αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου για τρεις εγκρίσεις ως τώρα Ξέρουμε ότι οι δύο τελευταίε θα περάσουν και στην Ολομέλεια την, επόμενη εβδομάδα. Ε, για τα του Ριτ τα έχουμε ξανασυζητήσει. Τώρα για το σχέδιο ψηφίσματος και τη διάρκεια αυτή τη ε, έγκριση. Ε, εδώ το σχέδιο ψηφίσματος αναγνωρίζει ότι πάνω από 400 ε, ε, σημεία παραγωγής και εργαζόμενοι επηρεάζονται από την συγκεκριμένη έγκριση και πόσο θα διαρκέσει. Πριν μπω σε λεπτομέρειες, να πω ότι αναστολή τη έγκριση σημαίνει ότι οι εταιρείε πρέπει να σταματήσουν να παρασκευάζουν και να χρησιμοποιούν τι ουσίε την επόμενη κιόλα λήψη τη απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από του εκατοντάδε χιλιάδε εργαζόμενοι μπορεί και να χάσουν τη δουλειά του. Η αλυσίδα παραγωγή ε, διακόπτεται και αναστατώνεται και θα υπάρξουν σοβαρέ οικονομικέ και κοινωνικέ συνέπειε μεταξύ άλλων σημεία παραγωγής που θα σταματήσουν να λειτουργούν και αποστολή της παραγωγής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα προϊόντα που έχουν τύχη επεξεργασίας με τριοξίδιο του χρώμιου δεν περιέχουν πια την ουσία και μπορούν ελεύθερα να τα εισάγουμε, ε, μπορούμε ελεύθερα να τα εισάγουμε από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε ε, δει χωρίς ιδιαίτερη προσοχή την αντίρρηση αυτή και τις εγκρίσεις. Έχουμε λάβει υπόψη όλες τις πτυχές που αναφέρει το ψήφισμα. Για παράδειγμα, αναρωτηθήκαμε αν η έγκριση πρέπει να περιοριστεί σε κράτη-μέλη ε, που θα αποφασίσει η Επιτροπή ΡΙΤΣ ε, πριν δοθεί. Η πρώτη αυτή συζήτηση που έγινε για εμά έδειξε ότι 27 από τα 28 κράτη-μέλη υποστηρίζουν ξεκάθαρα την πρόταση να δοθεί η έγκριση. Και αν δούμε το σχέδιο κειμένου που ε, χρησιμοποίησε ως βάση για να προβάλλει αντίρρηση η δική σας Επιτροπή. Ε, 24 από τους 28 ψήφισαν υπέρ στη δική μας Επιτροπή του ΡΙΤΣ. Οι χρήστε τη χρειάζονται αυτή την ουσία. Έχουμε κάνει λοιπόν διαφορετική ανάλυση και διαφορετικέ προσπάθειε να περιορίσουμε την ε, παροχή τη έγκριση και σε συγκεκριμένε χρήσει, ειδικά όταν είναι απολύτω απαραίτητη και όταν δεν υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ. Το σχέδιο ψηφίσματος το ίδιο αναγνωρίζει ότι χρειάζεται έγκριση για ορισμένους τελικούς χρήστες ε, στο τέλος της αλυσίδας παραγωγής και εκείνη ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν ξεχωριστή έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν ξεχωριστή έγκριση ή να έχει η Επιτροπή τη δυνατότητα να δώσει ε, εξατομικευμένα ή να αποσύρει την έγκριση. Αυτή τη στιγμή αναλύουμε την απόφαση του δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου και εκεί το Γενικό Δικαστήριο επέκρινε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή ΕΚΑΣ για τα θέματα αυτά που δεν μελέτησε επαρκώς τις δυνατότητες χρήσης εναλλακτικών όπως είχαν υποβληθεί στις πρώτερες διαβουλεύσεις. Και τελικά έδωσε την έγκριση. Όμω το δικαστήριο κατέστησε σαφέ ότι τέτοιου είδου ισχυρισμοί θα πρέπει να ε, τεκμηριώνονται στο πλαίσιο τη συγκεκριμένη έγκριση έχουμε αναλύσει διεξοδικώ όλε τι σχετικέ πληροφορίε. Και είδαμε και τι εναλλακτικέ τεχνολογικέ λύσει, τι λεγόμενε PDD. Οπότε Δώσαμε έγκριση για τη Λάνξες και για την ε, λεγόμενη έγκριση Γεχάντη με ρήτρα αναθεώρησης και μέγιστο όριο 7 χρόνια. Μέχρι εναλλακτικέ τεχνολογικές λύσεις να είναι έτοιμες και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αγορά πέραν της απόρρεψης της έγκρισης, η Επιτροπή προτείνει να χορηγείται η έγκριση για πολύ περιορισμένη διάρκεια και για πολύ περιορισμένο σύνολο χρήσεων. Με συγκεκριμένε αιτήσει αναέγκριση και πολύ αυστηρέ προποθέσει. Να θυμίσω ότι οι προποθέσει αυτέ έχουν να κάνουν με την ακριβή χρήση τη ουσία, 5 ως 20 φορές αυστηρότερες από τα όρια έκθεση για το χώρο εργασία και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το είπαν αυτό το Δεκέμβριο του 2017. Ε, εν είδη συμπεράσματο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι έχει βρει τη σωστή ισορροπία σε σχέση με το σχέδιο της αίτηση που καλύπτει πλήρως όλες τις ε, δυνατότητες άρνησης βάσει του κανονισμού Ρίτσα. Ευχαριστούμε κύριε Χόισλινγκ. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά τι μας λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, τα αναγνωρίζει και τα επιβεβαιώνει, αλλά δεν πιστεύω ότι βγάζετε τα σωστά συμπεράσματα από την απόφαση του δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου. Εγώ δεν βλέπω εδώ διάκριση με τη σημερινή περίπτωση που μας απασχολεί. Τώρα μπορούμε να ακούμε διάφορα επιχειρήματα και η κυρία Γκροστέτ λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτό που λέτε. Ότι αν το περιορίσουμε υπερβολικά θα παράγονται αυτά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι επιχείρημα είναι αυτό, ότι αν το απαγορεύσουμε εμείς θα τα βγάζουν οι άλλοι. Μα έχουμε μια σαφή νομοθεσία που λέγεται REACH για τα χημικά και θα πρέπει να την τηρούμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ γενναιόδορη στην ερμηνεία της νομοθεσίας REACH. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Και αναγνωρίζουμε στο ψήφισμα ότι υπάρχει διαφορά ε, ε, αν το επιτρέπω για τη διαστημική τεχνολογία ή για την επιχρωμίωση της θήκης του κραγιών. Δεν το καταλαβαίνετε ότι έχει διαφορά αυτό. Και θα πρέπει να ε, είναι διαφοροποιημένη η αδειοδότηση. Δεν το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι διαφώνησε και το Συμβούλιο και πολύ καλά έκανε. Ε, η Γερμανία το καταψήφισε ε, πράγμα που με εκπλήσει κατά τα άλλα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε άσπρο μαύρο ότι απειλούμε τη βιομηχανία στην Ευρώπη και είναι αυτό επιχείρημα. Ε, τότε να το καταργήσουμε το ρίτς αν δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την νομοθεσία που εμείς έχουμε εγκρίνει. Μήπως να το ξανακοιτάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την αναγκάσουμε να ε, πει ε, πολύ συγκεκριμένα ποιες είναι οι αλλακτικέ λύσεις και ε, πότε θα αδειοδοτείται το προϊόν όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση και υποκατάστατο, όχι γενικά. Γιατί καταργεί το ρίτσι στην ουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση και προχωρούμε στο επόμενο θέμα της μέρης της δέταξης που είναι οι ψηφοφορίες. They are announced to be at 10 so... Οι οποίες έχουν ανακοινωθεί για τις 10. Περιμένουμε λίγα λεπτά και να πάει 10 η ώρα και να έρθουν οι συνάδελφοι. Well, everyone. I invite you to... Λοιπόν, σας καλώ να πάρετε θέσεις για την ψηφοφορία. Λίγες είναι οι ψηφοφορίες ε, ηλεκτρονικές και δεν νομίζω να υπάρχουν και ιδιαίτερα ζητήματα. Ε, οπότε παρακαλώ να έχετε έτοιμες τις κάρτες σας. Είστε έτοιμοι υπέροχα. Λοιπόν, ψηφίζουμε πρώτα για την ε, προσωρινή συμφωνία που προκύπτει από τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός προγράμματος για το δράση για περιβάλλον και το κλίμα. Το πρόγραμμα LIFE δηλαδή. Άρχεται η ψηφοφορία. follow you. Okay. We have an... Πολύ ωραία. Υπάρχει μία αποχή από την κυρία Γιάρτε Μάκη. You said like this, so I thought it's an abstention. You vote... αποχή νόμιζα. Α, υπέρ. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το επόμενο κείμενο έχει να κάνει με την έγκριση ενός σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής για τον προπολογισμό 2020 και την σχετική εντολή για τον τρίλογο, τον τριμερή διάλογο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε για ένα μια έτσι ψηφίσματος για μια αντίρρηση σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση κάποιων ε, χρήσεων του τριοξιδίου του χρωμίου. Αυτή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Όμως, οι εργασίες μας συνεχίζουν. Κοινή ε, ακρόαση, δημόσια ακρόαση στις 10.30 με την Επιτροπή Στην 4Q1 θα γίνει αυτή η κοινή ακρόαση. Είναι η τελευταία μας ε, συνεδρίαση. 2 Απριλίου ακόμα ενδεχομένω θα έχουμε μία. Μαζί με την Επιτροπή Αναφορών είναι η ακρόαση